λαμβάνοντας πάντα βέβαια υπόψη την σωματική ε, ακαιρεότητα του προσωπικού μας και προσβλέπω στο ψήφισμα που, πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τα τελικά σας σχόλια. Έτσι τελειώνουμε το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τη δήλωση της υπασεκπροσώπου για την κατάσταση στη Συρία. ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο και πάλι στην υπατεκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δήλωσή της για τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, όλοι εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας από την τρομερή βία στη Συρία ε, οι δυνάμεις του καθεστώτος βομβάρδισαν πόλεις, ε, αμάχους, παιδιά. Εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα να σταματήσει η βία και η σκοτομή και όλοι ανησυχούν πάρα πολύ διότι υπάρχει το ενδεχόμενο της περαιτέρω στρατιωτικοποίησης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Η αυξημένη βία τις ε, μέρες μέχρι την προθεσμία στις 12 Απριλίου ήταν απαράδεκτη ε, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε σχέση με βομβαρδισμούς στην Όμσε, στην Χάμα και Ντέρα σκοτώθηκαν άμαχοι και αυτό είναι τρομερό. Ε, η βία έχει μειωθεί αλλά αυτό δεν αρκεί. Πάλι ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πιέσουμε για την άμεση πάυση της βίας για την εφαρμογή του σχεδίου ΑΝΑΝ. είναι πάρα πολύ ε, και ασταθής η κατάσταση. Ε, στην Χόμ, στην Άννα, στο Αλέπο ε, βλέπουμε τραγικά πράγματα. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ομόφωνα, ομόφωνα ε, τονίζω το Σάββατο ενέκρινε ψήφισμα για την άμεση ανάπτυξη μιας ομάδας 30 στρατιωτικών παρατηρητών στη Συρία για να αναφέρουν την εφαρμογή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός και της Βίας. Έφυγαν την Κυριακή για τη Συρία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη για την εφαρμογή του σχεδίου των έξι σημείων του Κόφη Ανάνα μαζί με τους προσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας και από τη φόρο τιμής ε, στη δουλειά και αφοσίωσή τους και όλα τα κράτη-μέλη δεν εφίστηκα προσπαθειών για να διασφαλίσω ότι η διεθνής κοινότητα θα μιλήσει με μία φωνή. Εγώ και οι υπηρεσίε μου ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τη Ρωσία και την Κίνα την περασμένη ε, φορά στα πλαίσια της συνάντησης ε, G8 στην Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τη θέση τους το ψήφινο του Συμβουλίου Ασφαλείας τέλος ε, είναι μια ε, ενιαία έκκληση από τη διεθνή κοινότητα προς το καθεστώς και παραθέτω ε, η κατεπίγουσα συνολική άμεση εφαρμογή από την κυβέρνηση της Συρίας όλων των στοιχείων της πρότασης του απεσταλμένου με τα έξι σημεία. δεν υπάρχει θέμα επιλογής, δεν είναι προαιρετική η πρόταση των έξι σημείων. Θα πρέπει να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση καθ' ολοκληρή θα πρέπει να ε, ε, αποσυρθούν τα στρατεύματα, ο βαρύς οπλισμός, ε, να μην βομβαρδίζουν τους φιλιρινικούς διαδηλωτές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια δημοκρατική μετάβαση στη Συρία η οποία θα ανταποκρίνεται στις νόμες, στα νομεοράματα όλων των Σύρων. Παρακολουθούμε από κοντά, έχουμε ε, ζητήσει από όλα τα μέρη να ε, συμφωνήσουν με το σχέδιο του, του Ανάν και βέβαια ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι το ψήφισμα είναι μια ευκαιρία ώστε το καθεστώς να αλλάξει η πορεία και να συνεργαστεί. Ε, εμείς από την αρχή θέλαμε ομόφωνη δράση και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να συνεχίσουν να στηρίζουν τον Κόφι Ανάν στις προσπάθειές του και να διασφαλίσουν να ε, γίνει λειτουργική μια αποστολή παρακολούθηση στη Συρία χωρίς καθυστέρηση. Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να συνεχίσουν να παίξουν, να παίζουν έναν κεντρικό ρόλο στην ε, επίτευξη της λύσης αυτής της σύγκρουσης ε, θα πρέπει να ασκήσουν την επιρροή τους. Επίσης, ξέφρασα την υποστήριξή μου στον ειδικό απεσταλμένο του Νανάν και του είπα και στο Γενικό Γραμματέα Μπανκιμούν που τον είδα χθε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα κάνουν ε, ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την ε, αποστολή αυτή παρακολούθηση. Ε, Εμεί ήδη προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε χώρο ε, βελτιωμένης επικοινωνίας και παρέχουμε επίσης και εκπαίδευση για να αναπτύξουμε την ανάλυση και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης. Επίσης την περασμένη εβδομάδα ε, συγκάλεσα την πλατφόρμα για την κρίση με όλες τις υπηρεσίες ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και την Επιτροπή. Επίσης σε συνεργασία έγινε καλός συντονισμός και με την κυρία Γεωργίεβα και ε, λάβαμε υπόψη μας και επικοινωνήσαμε όλες τις γειτονικές χώρες της Συρίας και τους πρεσβευτές της Βρυξέλλες. Επίσης συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική και σύντονη απόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εμείς ε, ε, ε, αναστήλαμε κάθε συνεργασία, διμερή συνεργασία, τη συμμετοχή της Συρίας σε περιφερειακά προγράμματα κλπ. Παρ' όλα αυτά διατηρήσαμε τη βοήθεια γιατί αυτή είναι προς όφελος του συριακού πληθυσμού των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αντιπολίτευση. Θα συνεχίσουν επίσης προγράμματα με τους φοιτητές ε, Επίση παρέχουμε στέγη, ε, φάρμακα, τρόφιμα, ό,τι χρειάζεται. Έχουμε ε, μια συμβολή με 29 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία και στις γειτονικές περιοχές. Επίσης είναι σημαντικό να στηρίξουμε και αυτές τις γειτονικές χώρες. Όταν πήγα στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών Νταβούτογλου ε, ο οποίος και θα, επίσης θα συνδεθεί με το ε, σχήμα αυτό της βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό. Η απόκριση της Τουρκίας ήταν εξαιρετική. γρήγορα, με επαγγελματισμό, ε, συνέβαλαν στην στήριξη 25.000 προσφύγων στο έδαφος τους πρόσφερα βοήθεια από εμά, τον Υπουργό Εξωτερικών τον Βούτογλου, ε, για οτιδήποτε χρειαστεί και παραμένω σε στενή επαφή μαζί του. Επίση, συνεργαζόμεθα στερνά με την Ιορδανία και τον Λίβανο και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά του. Αρχίσαμε επίση να συζητούμε τι λεπτομέρειε αυτή τη στήριξη με τον Υπουργό Εξωτερικών Νασέρ Τζουντέ. Είναι σημαντικό να δράσουμε γρήγορα, να συνδεθούμε ναι, στενά με τα επιτόπια Υπουργεία. Πολλοί εκτοπισμένοι ε, ζουν με τις οικογένειές τους, όχι σε καταβλισμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη υποστήριξη που θα συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη στις οικογένειες που τους υποδέχονται ε, και τους φιλοξενούν ε, υποστήριξη των περιοχών και των πληθυσμών που πλήττονται άμεσα από την εισρωή των σύρων. Ε, με τον ε, Επίτροπο ε, Φούλε θα συνεργαστούμε. Ήδη έχω προτείνει 23 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, γιατί από το μέσο γειτονία, ε, το οποίο είναι για την κοινωνία των πολιτών για τους πρόσφυγες και τους πληγέντες πληθυσμούς. Θέλω επίσης να πω ότι θα συνεχίσω με τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα στο βαθμό που η καταστολή συνεχίζεται. Ο τελευταίος γύρος των κυρώσεων εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών 23 Μαρτίου και ήδη τώρα δουλεύουμε πάνω σε μια νέα σειρά κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων σήμερα η ομάδα μου είναι στο Παρίσι και συμμετέχει ε, στην ομάδα εργασίας για κυρώσεις ε, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει η αντιπροσωπεία μας ανοιχτή στη Δαμασκό. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε ε, επιτόπου ένα μάτι και αυτή. Ο Συριακός πληθυσμός μας ζήτησε να μην φύγουμε. Επίσης έχουμε πολλούς διπλωμάτες κρατών μελών που αποφάσισαν να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους στη Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια και με, για τις επαφές μας με την, τις ομάδες αντιπολίτευσης στη Συρία πολύ σημαντικό αυτό και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ ιδιαίτερο ρόλο να παίξει. Σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να, και εσείς για να έρθουμε σε επαφή με τις ομάδες αντιπολίτευσης. Ο στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να δουλέψουν από κοινού προς καλύτερο συντονισμό, να συμφωνήσουν, να βρεθεί μια λύση που θα είναι χωρίς αποκλεισμούς, που θα είναι δημοκρατική λύση. Χρειάζεται κοινό όραμα για το μέλλον της Συρίας, όπου όλοι οι Σύροι, όλης κάθε προέλευση ε, ε, θα είναι ελεύθεροι και ίσοι. Επίσης η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα συνεχίσει να συναντάται με ομάδες αντιπολίτευσης ούτως ώστε να τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το μέλλον της Συρίας είναι στα χέρια του λαού της Συρίας. Η ζωή τους, τα δικαιώματά τους, τα οράματά τους θα πρέπει να τύχουν σεβασμού. Ε, το, ε, θα πρέπει ο πρόεδρος Ασάντε να ε, βάλει τα λόγια σε πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στο, στη Συρία παίζεται ένα τριπλό παιχνίδι. Καταρχήν ε, η επιρροή του Ιράν ή της Σαουδικής Αραβίας, ο ρόλος της Αραβικής Άνοιξης και επιπτώσεις, αλλά και ο ρόλος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών που ε, παραγωνίζονται περισσότερο από τον ανερχόμενο ρόλο της ε, Κίνας και της Ρωσίας. Είναι σημαντικό το σχέδιο και το ψήφισμα του ΟΗΕ. Θα πρέπει όμως η ψηφοφορία και η στάση αυτών των χωρών για την κατάσταση στη Συρία να είναι συμβατά. Η διπλωματική οδός είναι πιο αργή σε ό,τι αφορά την αλλαγή της κατάστασης. Θα πρέπει να στηρίξουμε όμως τους τοπικούς πληθυσμούς. Κυρία Άστον, θα πρέπει να στηρίξουμε το σχέδιο του Κόφιανάν Ανάν, αλλά σίγουρα φαίνεται να θέλουμε ένα διπλό μήνυμα στην διεθνή κοινότητα. Φενός, ο κύριος Ελασάντ ε, παραμένει στην εξουσία εδώ και καιρό ε, και γνωρίζει ότι με το βέτο της ε, Ρωσίας και της Κίνας συνεχίζει ατιμόρυτα να κατασφαγιάζει τον πληθυσμό του και Ταυτόχρονα θέλουμε ε, και το μήνυμα ότι βαρχιπρόθεσμα δεν διαφαίνονται λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν όλους αυτούς τους παράγοντες να τους σταθμίσουμε. Είναι αξιέπαινη η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ενίσχυση και την ε, κινητοποίηση των ε, κονδυλίων με την Αρμόδια Επιτροπή Γεωργίευα για να στηριχθεί η αποστολή μας εκεί. Αλλά όπως είπε και ένας στη χώρα μου, με βάση το, κόφι, το σχέδιο του Κόφι Ανάν, η επίλυση της σύγκρουσης θα πρέπει να ξεκινήσει ε, από τον Ασάτ και να ολοκληρωθεί με, την, ε, με το πέρας της ε, εξουσίας του. Κύριε Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαζί με την κυρία Γκομές πήγαμε στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου αρχές Απριλίου για να συναντήσουμε συγκεκριμένα ένα κομμάτι της Συριακής ε, ε, αντιπολίτευσης που είχε φτάσει μέχρι την Πυρητό, αλλά και για να καταλάβουμε καλύτερα τους κινδύνους για τον ε, Λίβανο από την ένταση τη γενικευμένη μεταξύ των και των Σιτών που θα προκληθεί από την σύγκρουση στην Συρία. Τι βγαίνει από όλα αυτά. Ε, δεν ξέρω αν έχω πιο ξεκάθαρες ιδέες από ό,τι στην αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει από όλα αυτά που ακούσαμε από τους Σύριους, ο φόβος ενός πολέμου εξαντανακλάσεως, ε, λόγω της γειτονίας δηλαδή, ε, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Σουνιτών και Σιτών στη Συρία, με ε, επέμβαση ενδεχομένω της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ κλπ. Όλο, αυτός ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Φαίνεται πραγματικά ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ είναι μία ε, πιθανή λύση πέραν του ε, φιλίου πολέμου στην Συρία. Δεν είναι εντελώς ικανοποιητική, αλλά αυτό είναι το αίσθημα που βλέπουμε να επικρατεί εκεί. Ένα σχέδιο ναν, αλλά ένα σχέδιο ναν βελτιωμένο, ε, λειτουργικό, που θα προέβλεπε την έξοδο του ΑΣΑΔ βραχυπρόθεσμα. Και για το σκοπό αυτό χρειάζονται ακόμα πολλές προσπάθειες και πρέπει να γίνουν συζητήσεις ε, με την Συριακή Αντιπολίτευση για να γίνει λειτουργικό το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αλλά ο φόβος ε, ε, φιλίου πολέμου είναι πραγματικά πολύ υπαρκτός. Δεύτερον, οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι πραγματικά μία ε, προτεραιότητα. Όχι μόνο ανθρωπιστική, αλλά πολιτική μέσα στο Λίβανο. Είναι μια πολιτική προτεραιότητα. Πρόκειται για αντιπολιτευόμενους της ε, Συρίας που ε, μπερδεύονται με τους Χεσμολά. Πρόκειται πραγματικά λοιπόν για μια πολιτική προτεραιότητα και τελειώνω. Ήθελα να σας πω κυρία Άστον πολύ σωστά διατηρήσατε μια πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δαμασκό. Κάντε όπως την Βεγγάζη. Διακόπτεται η κυρία. Λυπάμαι κύριε Ντεκάιζερ, αλλά έχετε υπερβεί κατά πολύ τον ε, χρόνο σας. Θα δώσω τώρα το λόγο για τρία λεπτά στον κύριο Φερχόφστα. Μην θυμώνετε κύριε Ντεκάιζερ, πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο και την τάξη εδώ πέρα. κύριος Φερχόφστατ. Κυρία Άστον, δώσατε μια πολύ, κάνατε μια πολύ διπλωματική ομιλία θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να σας πω, δεν συνηθίζω να συμφωνώ με τον κύριο Σαρκοζή, αλλά αυτή τη φορά ομολογώ ότι έχει δίκιο. Δεν πιστεύω ότι έχουμε πια σχέδιο ΑΝΑΝ ή ότι είναι λειτουργικό το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ας δούμε κατά πρόσωπο ε, τα γεγονότα. Έχουμε πάνω από 100 παραβιάσεις τις τελευταίες δύο μέρες του σχεδίου ΑΝΑΝ και ήδη είναι, τις έχουμε εντοπίσει. Πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν χθε τη ζωή τους. Δεν ξέρω πόσες ε, νεκρούς είχαμε σήμερα στη Σύρια. Πώς λοιπόν μπορείτε να μιλάτε για σχέδιο Ανάν, για ένα σχέδιο που δεν εφαρμόζεται στην πράξη από τον Μπασάρα Λασάντ. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνει η ευρωπαϊκή κοινότητα τι είναι, να περιμένει να σκοτωθούν εκατοντάδε χιλιάδες άνθρωποι πριν αναγνωρίσει η διεθνή κοινότητα ότι το σχέδιο Ανάν δεν λειτουργεί επειδή ο Μπασάρα Λασάντ δεν θέλει, δεν ε, είναι πρόθυμος να το εφαρμόσει. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν και πάλι σε μια κλιμάκωση των ε, ε, βιοπραγιών και των θανάτων στη Σύρια. Μιλήσαμε για παρατηρητέ τη Διεθνού Κοινότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ναι, να του υποστηρίξουμε. Ποιου να υποστηρίξουμε, να, για να δώσουμε 200, για να ε, ε, εγκαταστήσουμε εκεί 250 παρατηρητές χρειαζόμαστε χιλιάδες στρατιωτικούς ή αστυνομικούς να τους προστατεύουν να εξασφαλίσουν την ε, σωματική τους ασφάλεια όταν έχουμε 250 παρατηρητές στη Συρία πόσους στρατιώτες χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την προστασία τους αλλά ε, χρησιμοποιούμε τους στρατιώτες για να προστατεύσουμε τους δικούς μας παρατηρητές και όχι τους Σύριους που βρίσκονται στο έλεος του Μπασάρα Λασάντ. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι σωστός τρόπος για να συνεχίσουμε. Αυτό που θα πρέπει να διαπιστώσουμε κυρία Άστον είναι κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Ότι το σχέδιο Ανάν δεν λειτουργεί, ότι ο Μπασάρα Λασάντ συνεχίζει να σκοτώνει το λαό του, ότι ο Μπασάρα Λασάντ αθετεί τις υποσχέσεις του, ότι απλώς συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, τα γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα της παρατήρησης και της προστασίας των παρατηρητών. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αναλάβουμε δράση ε, ασφαλείς ζώνες, ανθρωπιστική διάδρομη και υποστήριξη της, της Συριακής Αντιπολίτευσης. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αν θα το κάνουμε με το Συμβούλιο Ασφαλείας, καλώς. Αν δεν γίνεται με το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαιτίας της θέσης της Ρωσίας και της Κίνας, ας το κάνουμε χωρίς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πάντως η διεθνής κοινότητα έχει υποχρέωση να δράσει. Και τέλος μια ερώτηση, κυρία Άστον. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το τελευταίο περιστατικό με ένα γερμανικό ε, πλοίο που προσπαθεί να παραδώσει όπλα στη Συρία και που καταστρατηγεί κατάφορα το εμπάργο όπλων. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το επεισόδιο. Όπως είπε η κυρία ε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σφυρί σας και να μας διακόπτετε όταν μιλούμε για τόσο σοβαρά προβλήματα όπως η κρίση στη Συρία. Κύριε Φερχόφστατ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρούμε τον κανονισμό και τις διατάξεις. Είχατε τρία λεπτά μπορείτε μόνο σας να κανονίσετε την κατανομή των σημείων, αλλά μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά. Κύριε Μπράντνερ. Κύριε Πατή, εκπρόσωπε, της, ε, αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάσταση είναι εφικτή και απαράδεκτη στη Συρία Πιο σημαντικό είναι να εξακολουθήσουν οι πιέσει ούτω ώστε αεροσκάφη, ελικόπτερα παρατηρητών και επιχειρήσει υποστήριξη ε, να μπορούν να κινηθούν. Γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα και πρέπει να υποστηρίξουμε πολιτικώ και οργανωτικώ την αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε του άλλου να του επι... υποστηρίζουν επιλεκτικά. Διότι έτσι έχουμε τον κίνδυνο να μην δημιουργηθεί ε, κοινή προσέγγιση. Ε, Αυτό είναι ο ρόλο μας ανθρωπιστικά τα δικαιώματα των προσφύγων θα πρέπει να τα εγγυηθούμε. Το να πυροβολούν τους πρόσφυγες από οποιαδήποτε πλευρά είναι απαράδεκτο. Τούτο λεχθέντος έχουμε και εμείς καθήκον να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες στι χώρε όπου καταφθάνουν και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σταματήσει η ματοχυσία στη Συρία και θα πρέπει να εφαρμόσουμε με αυστηρότητα το δικό μας εμπάργκο για τα όπλα. Δύο γεγονότα από 10 Ιανουαρίου οι κυπριακέ Αρχές επέτρεψαν να ανεφοδιαστεί ρωσικό σκάφο και να ελιμενιστεί ρωσικό σκάφο που είχε πάνω από 59 τόνου όπλα για τον Ασάντ παρά σαφή στοιχεία του επικινδύνου φορτίου που είχε και αυτό είναι εξωφρενικό και παράδεκτο. Κύπρο δεν μπορεί να ε, εξαγοράσει τα οικονομικά της προβλήματα από τη Ρωσία εις βάρος την πολίτηση της Συρίας. Και 13 Απριλίου ο γερμανικό σκάφος που είχε σημαία Αντίγκοα και Βαρμπούντα ε, σταματήθηκε καθοδόν προς Συρία. Άλλαξε φαίνεται πορεία το σκάφος αλλά σήμερα αγνοείται η θέση του ακριβή και αυτό είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι το εμπάργκο των όπλων ισχύει και εφαρμόζεται. Έχω στείλει ερώτημα με προτεραιότητα αυτό το θέμα και ζητώ να διαρευνηθεί ο ρόλο τη Κύπρου στο επεισόδιο που προανέφερα. Μέχρι τώρα δεν ε, μου δώσετε κάποιε πληροφορίε. Άρα είναι κατεπήγον και σας ζητούμε σε ανοιχτή επιστολή να διερευνήσετε αυτά τα γεγονότα και επιτέλους να υπάρξει πραγματική εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής του εμπάργου. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω προσωπικά αυτή την επιστολή και προσβλέπω στην απάντησή σας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν δέχεστε ε, κάποια ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Ο κ. Κασουλίδης. Έχετε το λόγο κ. Κασουλίδη. Yeah, Blue card, could you take... Είναι πρώτη για γαλάζια κάρτα. Θα την αποδεχτείτε. Όχι, ε, προσοχή, δεν είμαστε για φωτογράφηση. Συμπαθάτε με. Και παρακαλώ, βάλτε τα ακουστικά για να καταλάβετε αυτό που λέω για την γαλάζια κάρτα. Κασουλίδης, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι το καλοκαίρι μας πέρασε η Κύπρος ε, ε, χτυπήθηκε πάρα πολύ τρομερά διότι είχαμε αυτή την κατάσχεση των εκρηκτικών και αυτό αφορούσε την παραβίαση του εμπάργου όπλων προς τη Συρία, 14 νεκροί, οικονομικό ναυάγιο και επίσης επρόκειτο και για αυτό το οποίο μας αναφέρατε. Πρόκειται για αυτή την ε, εκδοχή που υποστηρίζει η κυβέρνηση της Νήσου. Είναι διαφορετική. Εγώ δεν έχω κανένα δισταγμό να καταδικάσω τη δική μου κυβέρνηση. Εάν η πάτη εκπρόσωπος η οποία παρίσταται μας ξεκαθαρίσει για το κατά πόσο πρώτο περί παραβιάσεως ε, διακόπτει ο Πρόεδρο. Δεν πρόκειται περί ερωτήσεω, δεν πρόκειται περί γαλάζια κάρτα. Σα ευχαριστούμε και διακόπτει τον κύριο Κασουλίδη. Yes, please. You have the floor. Έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Ξέρετε, όσον αφορά αυτό το εμπάργο των όπλων, ε, περιλαμβάνεται και το ότι δεν επιτρέπεται ούτε μεταφορά όπλων. Βέβαια, εξαρτάται για το πώς κανείς ορίζει τι θα πει διαμετακόμιση, μεταφορά. Όπως έγινε, είχαμε έναν εφοδιασμό, είχαμε τους Ρώσους που πέρασαν την Κύπρο. αυτό το οποίο θα σας πω είναι να γίνει μια έρευνα και έτσι να μάθουμε τις λεπτομέρειες, τα πραγματικά περιστατικά. Έρευνα. Και έτσι να μάθουμε τι είναι στην πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό να κάνει. Και έτσι να αποκτήσει αξιοπιστία σε αυτή την περιοχή. the second blue Ήθελα απλώ να ρωτήσω την συνάδελφο και νομίζω ότι θα δώσει κάποια πρόσθετη πληροφόρηση αυτό, εάν γνωρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη δια των δικηγόρων τη ασκήσει διαδικασία εναντίον της εταιρεία που μετέφερε τον συγκεκριμένο πλεισμό στην Συρία και αν αυτό κατά τη δική σας κρίση αποδεικνύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει επίσης να διερευνήσει αυτό το ζήτημα και το δεύτερο ερώτημα είναι αν γνωρίζετε γιατί η Κύπρος δεν είναι μέλος του Ασενάρ Arrangement, δεν το επιτρέπει η Τουρκία, και εάν ήταν, ε, τι περισσότερη πληροφόρηση νομίζετε ότι υποχρεωτικά των πραγμάτων θα είχε ε, για να μην καταλήξουμε στο αποτέλεσμα το οποίο εσείς καταγγέλλετε. Οπότε. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι τότε θεωρούσαμε ότι το πλοίο βρίσκεται στον λιμάνι και δεν το είχαν σταματήσει. Με 59 τόνους όπλων. Πώς είναι να το κάνει αυτό που θα πάει στον Άσαντ και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνει αυτό το όπλο. Οπότε τώρα ξέρουμε ότι κάτι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, ούτε βεβαίως είχαμε. Αλλά νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνομιλήσει με την κυβερνητική κυβέρνηση και τελικά να ανακαλύψουμε ότι ενδεχομένως όλα πήγαν πρίμα. Όμως θα πρέπει να γίνει αυτή η έρευνα, αλλιώς δεν μπορούμε να σιωπούμε. Ευχαριστώ. Και τώρα. Έχετε το λόγο κύριε Καρύμ για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπάτη εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε για το πόσο προσεκτικά διατυπώσατε τα της δηλώσεως σας σήμερα και καταλαβαίνουμε ποιες δυναμικές πρέπει να εξορροπήσετε σε σχέση με τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Συρίας που πρόκειται για μια φράση που την επικαλέστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί Ευρωπαίοι για και τις τελευταίες μέρες. Όμως το γεγονός είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε μια τέτοια κατάσταση μετασχηματισμού χωρίς να υπάρχει το, η μεταβλητή σημαντική της Συριακής Αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο τώρα λείπει. Ούτε έχω κανένα τους πληροφορία για το τι κάνει η διεθνής κοινότητα ή εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε ούτω ώστε να μπει στο παιχνίδι και η αντιπολίτευση. Επίσης, να σας πω αυτό το είπαμε και προηγουμένως, όσον αφορά με αυτούς τους ε, ακτιβιστές του Ιντερνετ για το ότι το καθεστώς με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, με πολύ καλό σχεδιασμό, με πολύ προχωρημένους τεχνολογικά τρόπους, τους επισημαίνει, τους συλλαμβάνει, τους φημώνει, δεν περνά το μήνυμα όσον αφορά τις αγριότητες που εκεί λαμβάνουν χώρα. στη συνέχεια για ένα λεπτό κύριος Μπέρντερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μία αποστρατιωτικοποίηση στη σύραξη στη Συρία είναι αναγκαία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πολιτική λύση του πρόβληματος. Το πρόβλημα όμω είναι ότι από γειτονικά κράτη εισραίουν πολλά όπλα στη Συρία. Μπορεί ίσω προληπτικά να δράσει η Ευρώπη στον Κολάν της Συρίας και στο νότιο Λίβανο υπάρχουν χιλιάδες κιανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών εκεί. Πολλοί από αυτούς έχουν και ευρωπαϊκή υπηκότητα. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, ένα μέρος αυτών των κυανόκρανων, Ευρωπαίων κυανόκρανων, δεν θα μπορούσε προσωρινά να τοποθετηθεί στα συριακά λιβανικά σύνορα, ώστε να γίνονται έλεγχοι εκεί ή στα συριακά ιορδανικά σύνορα. Δεύτερη ερώτηση. Μετά από την πίεση στις Συριακές αρχές, ασκείται τώρα πίεση στο Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας για να υπάρξει κάποια συμφωνία και λύση διότι χαιρετίζουμε το, το σχέδιο του Κόφι Ανάν. Σας ευχαριστώ και στη συνέχεια τηρήσατε το χρόνο σας. Και τώρα στη συνέχεια κύριος Χατζηγεωργίου παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μας να παρακολουθεί με απάθεια σφαγές που γίνονται εναντίον πολιτών σε κράτη της περιοχής μας και μάλιστα όταν οι σφαγές αυτές καθοδηγούνται από τους ηγέτες αυτών των κρατών. Νομίζω όμως παράλληλα ότι είναι σωστό να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα και να τα βάλουμε στην ισορροπία ή στην ζυγαριά. Πόσους χιλιάδες νεκρούς θα πρέπει να βάλουμε στη μια ζυγαριά για να δεχτούμε ότι αυτό αντισταθμίζει με μια αμφιλεγόμενη δημοκρατία που θα έρθει στη συνέχεια δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί σε αυτή την αίθουσα που να πιστεύουν ότι οι πενήντα μπορεί να κάνω λάθο και να είναι περισσότεροι χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε νεκροί στο ιράκ αντισταθμίζει το γεγονό ότι υπάρχει σήμερα στο ιράκ αυτό που ονόμασα πριν μια αμφιλεγόμενη δημοκρατία. πρέπει να στηρίξουμε την άποψη καμία εισαγωγή οπλισμού στην συρία από οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε διάδρομο και θα πρέπει να στηρίξουμε το σχέδιο ανάν χωρίς να δεχτούμε καμιά παραβίασή του για την περίπτωση της Συρίας. Είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε ποιο είναι το βάρος που παίζει η Συρία στην περιοχή και δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση ότι δεν πρέπει κανείς να λάβει υπόψη τη Συρία ή την Κίνα. Είτε το θέλουμε είτε όχι υπάρχουν οι γεωστρατηγικές συμπεριφορές των κρατών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και εμάς αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι το αποτέλεσμα να μην πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των νεκρών που υπάρχει σήμερα στη συρία. εάν αποκλειστεί η δυνατότητα να μπορούν να εισάγονται όπλα στη συρία μαζί με την επιμονή μας ότι το σχέδιο ανάν για τη συρία πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως είναι ο μόνος τρόπος να συγκρατήσουμε τα πράγματα και την αιματοχυσία. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Um, uh, from the visit uh, that, uh, De ε, από την επίσκεψη που έκανα η κυρία Ντεκάζερ και εγώ που πήγαμε στην περιοχή στο Βόρειο Λίβανο και θα είμαι σε επαφή με Σύριους πρόσφυγες και από άλλες επαφές είναι πέρανα ότι πράγματι υπάρχουν δύο πόλεμοι που λαμβάνουν χώρα. Λοιπόν, Νέα Υόρκη μεταξύ Ρωσίας, ΙΠΑ και Κίνας και επιτόπιος πόλεμος Σουνίτες υποστηριγμένοι από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία εναντίον Σιητών που υποστηρίζονται από το Ιράν που υποστηρίζει το καθεστώς Ασάντ. Μεγάλη υποκρισία και πολύ ανησυχητική. Συμπεραμβάνονται και τα κάτι μέλη. Μιλούσαν για ανθρωπιστικό διάδρομο και δεν κάνουν τίποτα κάτι μέλη γι' αυτό να υλοποιηθεί. Αυτό απαιτεί στατό, ασφάλεια για να υπάρχει ανθρωπιστικός διάδρομος. Όπου και αν ανοίξει. Στην Τουρκία, Φερρυπίν. Παίζεται ένα παιχνίδι πολιτικής υποκρισίας εκεί. Και απαράδεκτη παραβίαση του εμπάρκο. Αυτοί που αναφέρθηκε πάντα ευκρινιστούν αυτά τα επεισόδια από το κράτη-μέλη. Κρίσιμο την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει το σχέδιο Ανάν. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να αποφευθεί παρατεταμένος εμφύλιος πόλεμος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι ξεκάθαρο κάτι που δεν είναι στο σχέδιο Ανάν, αλλά πρέπει να είναι σαφές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε ο Ασάντ να φύγει από την εξουσία και θα πρέπει να πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αυτός και άλλα μέλη του καθεστώτος του για εγκλήματα κατά του λαού του Συρίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε το σχέδιο Ανάν, είναι πολύ σημαντικό, κυρίως όσον αφορά για την ασφάλεια των παρατηρητών, αν πρόκειται να πάνε εκεί οι παρατηρητές, όσον αφορά αυτές πτυχές. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες. Όχι μόνο αυτούς που είναι στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως το Λίβανο, που ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και να υποστηρίξουμε και τον πληθυσμό. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη Συριακή Αντιπολίτευση, ώστε να ενωμένει επί μιας δημοκρατικής ενιαίας πλατφόρμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα. Ο κύριος Ντεόφερ, παρακαλώ. Είναι θλιβερό και ντροπιαστικό αυτό το οποίο υφίστανται οι Σύριοι. Ω διαμεσολαβητή έκανε ο Κόφη Ανάν ό,τι μπορούσε αλλά φτάνουν αυτά όχι. Εφόσον η παγκόσμια κοινότητα, ιδιαίτερα η Κίνα και η Ρωσία δεν καθιστούν σαφέ στον Ασάντ ότι πρέπει να αποχωρήσει διότι η συμμορία του και ο ίδιο δεν μπορούν να αφήσουν την ειρήνη να ανθίσει εφόσον δεν φεύγει ο Ασάντ θα συνεχίσει να δολοφονεί του πολίτε του και δεν θα σταματήσουν οι δολοφονίες. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Όποιος νομίζει ότι με τον ε, Ασάντ και τους δίμιους του μπορεί να διαπραγματευτεί, αυταπατάται. Λίγη ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα για να μπορέσω να παρέμβω θα ήθελα να μπορέσω να μιλήσω χωρίς να με ενοχλεί αυτός ο θόρυβος. Όποιος νομίζει ότι με τον Ασάτ και τους δίμιους του μπορεί να διαπραγματευτεί με αυτούς, αυτά πατάτε. <clears throat> Έχει απόλυτο δίκιο όταν ζητείτε υποστήριξη για τους πρόσφυγες στα σύνορα μέχρι και την διάνοιξη ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου. Διότι όταν έχουμε εδώ μπροστά μας αυτή την κατάσταση πρέπει με ε, την βία να προσπαθήσει να πετύχει κάτι. Κανείς δεν θέλει κλιμάκωση της βίας αλλά δεν μπορούμε να είμαστε θεατέ. Πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα αναδίπλωση, ένα πρόγραμμα Β, Plan B. Βλέπω δυστυχώ όμω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η διαδικασία απόσπαση προσοχή του Προέδρου, ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Έχουμε πολλού ομιλητέ, επτά. Η κυρία Κρετού είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το πρόγραμμα σχέδιο Ανάν ήταν η τελευταία προσπάθεια να επιληθεί με ειρηνικό τρόπο η σύραξη στη Συρία. Όπως αναφέρθηκε, πάνω από 11.000 είναι τα θύματα της βίας στη Συρία. Χιλιάδες παραπάνω τραυματίστηκαν, άλλοι συνελήφθησαν παράνομα, άλλοι βασανίστηκαν. Όλες οι κυρώσεις δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και η εύθραυστη εκεχηρία η οποία έχει κατάφορα παραβιαστεί δείχνει ότι το καθεστώς του Ασάντ δεν είναι καθόλου καθόλου έντιμο όσον αφορά την παγκόσμια κοινότητα. Το καθεστώς της Δαμασκού μόνο στα λόγια υποτίθεται ότι συμμορφωνόταν ότι θα σταματούσε η βία. Όμως κλιμάκωσε τη βία. Παρότι δεν έχει επιτευχθεί λύση από το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουμε τη δήλωση της 31ης Μαρτίου που υποστηρίζει το πρόγραμμα του Αραβικού Συνδέσμου και του ΟΗΕ. Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που πρέπει να γίνει υπό τους όρους και παρουσία των εκπροσώπων του ΟΗΕ. Ευχαριστώ κύριο Στάνοξ στη συνέχεια Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική κατάσταση Συρία εξακολουθεί να επιδεινώνεται δυστυχώ. Σήμερα το απόγευμα είδαμε ότι οι συνδυνάμει Συριακή κυβερνήσεω ξεκίνησαν εκ νέου να βομβαρδίζουν την, τον ελεύθερο Συριακό στρατό και περιοχέ γύρω από το Χόλμ και έσπασαν την εκεχηρία που είχε εφαρμοστεί σύμφωνα με το σχέδιο ανάγκη του ΗΠΑ. Καλό την είπατε εκπρόσωπο να αναδιπλασιάσει τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τη πραγματευσίε τη διεθνή. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να, υπάρξει, να παρατητέ του ΟΗΕ να ξεκινήσουν γρήγορα τη δουλειά του και χωρί εμπόδια. Είναι σαφέ ότι Ασάντ έχει χάσει η αδίποτε μορφή ηθική κύρου για να μπορεί να κυβερνήσει τη Συρία σαν πρόεδρο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι αδίστακτε επιθέσει του άφησαν περίπου 9.000 πολίτε νεκρού ή τραυματίε. Η Συριακή κυβέρνηση θα πρέπει τελικά να αναλάβει τι ευθύνε για όλε τι δράσει τη και αν έχει παραβιάσει τι υποχρεώσει που είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, τότε θα πρέπει γρήγορα να επιβληθούν κυρώσει από όλη την διεθνή κοινότητα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πάσκα είναι ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι υπατή εκπρόσωποι. Ένα επιπλέον κράτος η Συρία στον αραβικό κόσμο όπου έχουμε αυτή την έκρηξη βίας και τη σύραξη έχουμε θύματα, χιλιάδες θύματα από πλευράς καταπίεσης του καθεστώτος, κυρίως άμαχους το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίε, να σταματήσει η βία και ο ίδιος ο Κόφι Ανάν με επιτυχία κατέβαλε προσπάθειες ε, ώστε να πιστούν οι εμπλεκόμενοι να δεχθούν το πρόγραμμα των έξι σημείων ώστε με τον τρόπο αυτό από πλευρά Ηνωμένων Εθνών να συνεισφέρει ο ΙΕ υπέρ τη Ειρηνή. Τώρα μέλη της, ε, παρατηρητές μπορούν να αποσταλούν, μπορούν να βρίσκονται στη Συρία σε διάφορες ε, τοποθεσίες ώστε να παρατηρήσουν, να υποπτεύσουν την τήρηση αυτού του προγράμματος σχεδίου εκεχηρίας ε, και να το εποπτεύουν η ε, οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν μπορεί να συνεισφέρει με κανένα τρόπο λοιπόν υπέρ της ειρήνης. Ο κύριος Όμπερμαϊερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σε σχέση με την Συρία έχει ένα οπλοστάσιο χιλιάδων πυράβλων και δηλητηριωδών αερίων πράγμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Ευρώπη επειδή η εμβέλεια αυτών των πυράβλων μπορεί να πλήξει την Ευρώπη. Δημιουργείται εδώ λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να συνεισφέρουμε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης εκεί. Πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος η ειρήνη. Η ειρήνη που πρέπει να αποκατασταθεί σε αυτή την περιοχή και να υπάρχει ένα ε, μετριοπαθέ καθεστώ, το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και τα δικαιώματα των μειονοτήτων κυρίως και των Κούρδων. Πρέπει ιδιαίτερα η Τουρκία να συνεισφέρει. Η Άγκυρα έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν να ε, συνεισφέρει περισσότερο. Πώς μπορεί λοιπόν να συνεισφέρει η Τουρκία και να μπορέσει η κατάσταση αυτή να σταθεροποιηθεί. Είναι σαφές ότι με την Τουρκία και την Συρία υπάρχει μια αιστεία σύραξης που μπορεί να απειλήσει και την ίδια την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής η κυρία Ζούμπε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο λαός της Συρίας θέλει περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη δικαιοσύνη επί πολλά χρόνια βρισκόταν ε, ε, το αίτημα αυτό έναντι της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι παρά η ε, κατατρόπωση, η καταπίεση των αμάχων και των αντιφρονούντων. Είναι εδώ ένα, μια σύραξη που από το εξωτερικό χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση, μισθοφόροι, τρομοκράτες που χρηματοδοτούν από το εξωτερικό για να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μια εσωτερική σύραξη της Συρίας αλλά μια πράξη αποσταθεροποίησης υπεριαλιστική ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τους πόρους αυτής της χώρας στη Μέση Ανατολή. Είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε μέσω του εθνικού διαλόγου που θα επιτευχθεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ ΕΕ και άλλες χώρες να μην αγνοούν τον ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίσουν οι αρχές ε, για να συνεισφέρουν υπέρ της ε, ε κατάπαυσης της ε, σύραξης. Ευχαριστώ. Thank you very much. And the last... Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μέλτσερ είναι τελευταίος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ως γνωστόν κατηγορεί η μία πλευρά την άλλη για τις ε, βιαιότητες και για το ότι υπήρξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτά σίγουρα δυσχεραίνεται η εφαρμογή του προγράμματος του σχεδίου ΑΝΑΝ με τα έξι ε, σημεία. Τώρα, αν μπορεί ο ΙΕ να συνεισφέρει ώστε η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση να διαπραγματευτούν ή αν πρόκειται απλά και μόνο για κάποια παραπλανητική κίνηση από πλευρά των εμπλεκομένων, σίγουρα θα αποδειχθεί τι τις επόμενες ημέρες και με τις ενέργειες του Αραβικού Συνδέσμου. Αν η αποστολή Ανάν δεν δώσει την ε, ευκταία επιτυχία πρέπει να αυξηθεί η πίεση από πλευράς μας. Όμως μια ε, άμεση επέμβαση όπως ζητούν ε, οι αντιπολιτευόμενοι με τη θέσπιση μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη Συρία δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει εδώ να μπορέσουμε να μάθουμε από τα σφάλματα που έγιναν στο παρελθόν με τη Λιβύη και να αποφύγουμε τέτοια σφάλματα στη Συρία. Σας ευχαριστώ και για τις τελικές παρατηρήσεις θα ήθελα να δώσω στον λόγο στην Βαρονέσα Αστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανέστατο από όλε τι παρεμβάσει ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και μεγάλο πάθο που αισθάνονται τα μέλη του Κοινοβουλίου και αυτό αντικατοπτρίζεται σε κάθε συζήτηση που έχω με οποιονδήποτε που ενδιαφέρεται για το ε, δράμα και τη φρίκη που υπόσχεται ο Συριακός λαός. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, συναισθηματικά είναι πολύ ελκυστικό και δυστητικά να μιλάμε για δρόμους ασφαλείας, ασφαλείς τόπους, ε, ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η βία στη Συρία καλύπτει 180.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν είναι κάπου απομονωμένα, είναι παντού η βία. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ανησυχούν για οτιδήποτε θα ενέπλεκε τους στρατιωτικούς που θα υποστήριζαν τις εργασίες τους και πρέπει να σεβαστούμε, να ακούσουμε γιατί έχουν εμπειρία αυτοί οι φορείς. Πέραν αυτού το για να πάει κανείς να αναπτύξει δυνάμεις επιτόπου είναι τεράστια προσπάθεια και χωρίς απόφαση του ΟΗΕ να γίνει κάτι τέτοιο είναι τεράστια πρόκληση. Uh, uh, Πώς να το πω, περίπου έτσι. Είναι σημαντικότατο λοιπόν να αναγνωρίσουμε τι ακριβώς εκπροσωπούν αυτές οι ιδέες πρέπει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό που συζητάμε ακριβώς, ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Δεύτερον, ο ΙΕ δεν έχει επιβάλει εμπάργκο όπλων, διότι δεν επετέφθη στο Συμβούλιο ασφαλεία συμφωνία. Εμεί έχουμε εμπάργκο όπλων και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και συνεργαζόμαστε με την Κύπρο και με τη Γερμανία. Θέλουμε να βρούμε λεπτομέρειε, να διερευνήσουμε τι ακριβώ έγινε. Και θα απαντήσω δίνοντα ε, πληροφορίε μου δοθούν. Τρίτον, Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, συνεργαζόμενοι όσο πιο στενά γίνεται με όλου του άλλου, ούτω ώστε οι ομάδε αντιπολίτευση να ενωθούν. Στην τελευταία συζήτηση που είχαμε τον Κόφι Ανάν, το είχε υπόψη του. Ήταν μέρη του. Πώ να δημιουργηθεί μια αιγίδα, να υπάρξει κάποια συνεργασία ε, γύρω από ένα τραπέζι, ούτω ώστε να παραμερίσουν τι διαφορέ του και να καταλήξουμε μια κοινή θέση. Και στην Κωνσταντινούπολη αυτό είναι τα βασικά θέματα. Εξακολουθούμε να συνομιλούμε με αυτούς και με τους συναδέλφους μας όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ενότητα της αντιπολιτεύσεως. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε επί του σχεδίου ΑΝΑΝ με τα έξι σημεία. Έχουμε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που μπορούμε να υποστηρίξουμε και όλοι να υπομισθούν τις ευθύνες τους. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Στη Συρία όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου και την κεχηρία κατάποση του πυρό και οι παρατηρητέ είναι έτοιμοι να εργαστούν και πρέπει να του υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να εργαστούμε όσο πιο σκληρά γίνεται, ώστε και τα έξι σημεία να εφαρμοστούν και να κάνουμε αυτό που μα ζήτησε ο Κόφη Ανάν. Να του προσφέρουμε την πλήρη μα υποστήριξη. Έχει τη δική μου υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρίε και κύριοι, η συζήτηση υπερατώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 12. Ε, Επόμενο σημείο προς συζήτηση είναι η κατάσταση στη Βυρμανία. Θα ήθελα να σας ζητήσω